Και όπως τονίστηκε στην Μαδρίτη στις 17 Σεπτεμβρίου, η αδίποτε λύση θα πρέπει να βρίσκει σύμφωνη και την Λιβύα. Και έχουμε τώρα κάθε μορφή επέμβασης διεθνούς που θα πρέπει να απορρευτούν. Και ούτε μπορεί να επιδέχεται αυτή η κρίση στρατιωτική λύση. Θα πρέπει ο εθνικός διάλογος να συμπεριλάβει τους πάντες. Επίσης θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο συντονισμός από όλους τους εμπλεκομένους για να πετύχουμε το στόχο μας. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα πρέπει να εστιαστεί στο πώς θα βοηθήσει τις προσπάθειες του Άντσιμιλ. Χρειαζόμαστε πρακτική ε, στήριξη των όσων γίνονται εκεί Χρειάζεται συντονισμός ε, της πολιτικής, των πολιτικών επαφών σε υψηλότερο επίπεδο με τους, θετικούς, ε, τους τοπικούς ε, παράγοντες όπως στη Μαδρίτη είχαμε επίσης και τις συναντήσεις στο πλαίσιο του άγγελου που οργάνωσε ο ΙΕ και η πολιτείε. Και έτσι θα πρέπει όλοι αυτοί οι τοπικοί παράγοντες, όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι να λυθούν, να βρεθεί μια λύση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιε κυρώσει κατά αυτόν που απειλούν την ειρήνη, που θέτουν ει κίνδυνο την τόσο δύσκολη υπόθεση του μετασχηματισμού του, της Λιβύης. Ο ΙΕΚ έχει ένα ψήφισμα σε σχέση με αυτές τις κυρώσεις, οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε το πώς αντέδρασε στο προηγούμενο καθεστώς οι διεθνείς κοινότητες. Και ήδη τόνισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η πρώτη προτεραιότητα και για τη Λιβύη αλλά και για τη διεθνή κοινότητα είναι το να μπορέσουμε να πετύχουμε μια κατάπαυση πυρός από όλες τις πλευρές και έτσι να έχουμε ένα πολιτικό διάλογο που να τους καλύπτει όλους. Ο ε, Άνσμιλ ε, στις 29 Σεπτεμβρίου κάλεσε τους πάντες να κάτσουν γύρω από το τραπέζι των ε, συζητήσεων, Ούτω ώστε να υπάρξουν κάποιοι βασικοί κανόνες και έτσι να ξεκινήσει πάλι μια διερεύνηση πολιτικής λύσης. Βέβαια, οι λεπτομέρειες ακόμα δεν έχουν καθοριστεί για αυτή τη συνάντηση. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ είναι έτοιμη να συμβάλλει και να βοηθήσει σε αυτή την διαδικασία που θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία και έτσι να συνεχιστεί ο μετασχηματισμός στη χώρα. Αυτό είναι η πρώτη, η κορυφαία μας προτεραιότητα. Να πετύχουμε την ε, ανακοχή, την κατάβαση πυρός και να μαζέψουμε όλους τους εμπλεκομένους γύρω από ένα τραπέζι συζητήσεων και να τεθούν κάποιοι βασικοί κανόνες. Όχι στη βία, όχι στην ε, εξωτερική επέμβαση και να έχουμε τις προϋποθέσεις τόσο ώστε η ίδια η Λιβύη να συνεχίσει την, ε, το μετασχηματισμό της αλλαγές και να συμμετάσχουν εκεί όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες της χώρας. Και αυτή είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα και σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Would like to ask now Mr. John Παρακαλώ τον κύριο Ζαν Ροκ που είναι επικεφαλής της μονάδας για την Αραβική Χερσόνησο, το Ιράν και το Ιράκ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. τα γεγονότα των τελευταίων 48 ώρων ήταν δραματικά. Πάνω από 100.000 ε, ε, Κούρδοι ε, έφτασαν στα τουρκικά σύνορα. Είχαμε ε, βομβαρδισμούς ε, με επικεφαλής των ΗΠΑ ε, στην Σύρια, αλλά πρέπει να σας πω πρώτον ότι ήδη είμαστε από καιρό προετοιμασμένοι για να πολεμήσουμε αυτή την πληγή του ε, ISIS ε, και ότι ε, γίνεται προσπάθεια να συμβάλλουμε στην επίλυση της κρίσης στη Συρία και στο Ιράκ. Πρώτα απ' όλα η κρίση στις χώρες αυτές ε, έχει κάποια κοινά στοιχεία, ε, πρώτο μεταξύ των οποίων ε, η ίδια η ISIS, αλλά έχουν οι δύο χώρες αυτές και πολλές διαφορές και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας προετοιμαζόμενοι για την ανταπόκριση μας σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως μπορούμε να αναφερθούμε σε πέντε κατηγορίες όσον αφορά την ανταπόκριση μας. Πρώτον, πιστεύω ότι πρέπει ε, να απομονώσουμε την ISIS, ε, να αποκόψουμε οποιαδήποτε πρόσβασή της σε χρηματοδότηση και σε οπλισμό και επίσης ε, να σταματήσουμε ε, τους ξένους μαχητές ε, που πηγαίνουν να πολεμήσουν με την ISIS. Θα πρέπει να σταματήσουμε την πρόσβαση δηλαδή νέων τζιχαντιστών στα προς, προς εκεί που βρίσκεται η ISIS αλλά και προς τις χώρες μας. Κοιτάξτε, τα σύνορα σε αυτή την πλευρά του κόσμου είναι ιδιαίτερα περατά ε, και ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο λαθρεμπόριο που βεβαίως είναι πηγή ε, ε, εσόδων για την ISIS έχει ξεκινήσει δε εδώ και πολύ καιρό. Δεν έγινε ξαφνικά όλη αυτή η διαδικασία ούτε την εφήβραν οι ίδιοι, απλώς τη χρησιμοποίησαν. Δεν είναι και πολύ εύκολο να το αντιμετωπίσουμε αυτόν γιατί οι κυρώσεις μας δεν είναι στοχευμένες ε, για να αντιμετωπίζουν μικρούς εμπόρους ε, οι οποίοι ε, περνάνε ας πούμε κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου από την Συρία ή από το Ιράκ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, εμείς προσπαθούμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα κορδόν σανιτέρ, έναν αποκλεισμό υγειονομικό κατά κάποιο τρόπο ε, στην εμπόλεμη περιοχή, ε, στο Ιράκ και αυτό το κάνουμε με την διεθνή υποστήριξη που υπάρχει στο ε, Ιράκ και τώρα ε, και στην Συρία. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει τις τελευταίες ε, ημέρες καταδεικνύει τη δυσκολία της καταπολέμησης του ISIS από ένα και μόνο μέτωπο. Ε, τους ε, σπρώχνουμε προς το βορειοδυτικό ε, Ιράκ, αλλά αυτό προκαλεί μεγάλα κύματα προσφύγων και στην Συρία και αυτό ακριβώς καταδεικνύει τη δύναμη που έχει η ISIS να αποσύρεται από πεδία μαχών στα οποία δέχεται επίθεση και να πηγαίνει πλέον προς άλλες κατευθύνσεις. Η δυσκολία της, στην ε, στρατιωτική ανταπόκριση, τουλάχιστον στο Ιράκ, όπου έχουμε κυβέρνηση φιλική ε, και που έχει ζητήσει ρητά την βοήθειά μας, πράγμα που δεν συμβαίνει στην Συρία, ε, γιατί το καθεστώς δεν είναι φιλικά προσκύμενο και δεν είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ξέρουμε πώς έχει κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ε, ξέρουμε όσον αφορά την αγορά των όπλων, ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα στο, ε, στους Κούρδους και στο Κουρδιστάν. Είπα, αναφέρθηκα ήδη σε δύο θέματα. Υπάρχει βεβαίως ε, και η πολιτική ε, απάντηση. Ε, ξέρουμε ότι έχει περιθωριοποιηθεί το ΙΖΙΣ στην κοινότητα των Σουνιτών του Ιράκ και η νέα κυβέρνηση γνωρίζει ε, και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά ε, το πρόβλημα έτσι ώστε ε, να ανακουφίσει τον φόβο τον οποίο έχει αναπτύξει πλέον ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τώρα έχουμε έναν νέο υπουργό ορισμό, έναν υπουργό εσωτερικών συγγνώμη, ε, θα δούμε ποιος θα είναι ο νέος Υπουργός Εσωτερικών ε, έτσι ώστε ε, να προχωρήσουν τα πράγματα στο μέλλον καλύτερα και περιμένει και η κοινή γνώμη του Ιράκ με μεγάλη αγωνία ποιος θα είναι ο νέος Υπουργός. Δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι για τους Σουνίτες και τους ηγέτες τους ενδεχομένως ορισμένες φορές να έχουν μια τακτική συνεργασία με τους με την ISIS, αλλά όσον αφορά την κυβέρνηση, ε, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να ρυθμιστεί η κατάσταση. Υπάρχουν φυσικοί αλλά και πολιτικοί κίνδυνοι για όσους προσπαθήσουν την προσέγγιση. Τέλος να θυμίσω ότι η συνεργασία με τους ε, τοπικούς περιφερειακούς εταίρους είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε ε, να μην θεωρηθεί η όποια κίνησή μας ή παρέμβασή μας ε, σαν μια προσπάθεια να καπελώσει η Δύση την Ανατολή ή αυτές τις περιοχές. Επίσης μιλισμονούμε ότι έχουν και αυτοί τη δικιά τους ατζέντα και τις δικές τους προτεραιότητες. Υπάρχουν Επίσης ε, ε, πολλές ε, τοπικές εντάσεις, ας πούμε Σαουδική Αραβία με Ιράν, Συρία με Τουρκία και θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια προσπάθεια συνολικής υπερκέρασης αυτών των τριβών έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα κοινό μέτωπο. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ενδεχόμενα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις συνάδελφοι, πολύ σύντομα παρακαλώ. Νομίζω ότι τη, συνάντηση, τη συζήτηση αυτή μπορούμε να την ε, συνεχίσουμε στις 3 η ώρα που θα συζητήσουμε για τη Γάζα. Θα βρούμε κάποιο χρόνο και γι' αυτό. Σε 10 λεπτά πρέπει να είμαστε στην ε, άλλη επιτροπή. Ο, κύριος είναι, ο πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριος Ντονζόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλουμε να απομονώσουμε αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση, το Ισλαμικό κράτος, κατά της οποίας σήμερα έχει δημιουργηθεί μια στρατιωτική συμμαχία. Πολύ καλό αυτό, συμφωνώ, επί της αρχής κανένα πρόβλημα. Αλλά τι θα γίνει με τις άλλες ομάδες. Γιατί αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι ότι και οι άλλες ε, τρομοκρατικές ομάδες, για παράδειγμα το μέτωπο Αλνούσρα και οι τελευταίες επιθέσεις στο Λίβανο, έχουν γίνει διάφορες ε, επιδρομές στο Λίβανο, έχουν γίνει απαγωγές και εκτελέσεις Λιβανέζων στρατιωτών, α, όχι από το Ισλαμικό κράτος, αλλά από το Αλνούσρα. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τα ΜΜΕ κυρίως ασχολούνται με το Ισλαμικό κράτος, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Ιράκ και ιδιαίτερο στη Συρία υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα έλεγα ότι είναι εξίσου επικίνδυνες. Η Αλνούστρα επίσης έχει μια στραγική διεθνιστική πολύ πιο σαφή από ότι το Ισλαμικό κράτος. Δεύτερον, μιλήσατε για τη συνεργασία με τα κράτη της περιοχής βεβαίως, ουσιώδες, θεμελιώδες. Αλλά εξακολουθώ να διερωτώ με τι ρόλο παίζει η Τουρκία, υποψήφια χώρα. Ξέρω τώρα ότι διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους ε, είναι σε χαόδη κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά, όλα τα υποψήφια κράτη έχουν κάποιε υποχρεώσει ε, σε θέματα εξωτερική πολιτική. Πρέπει να συγκλίνει η εξωτερική του πολιτική με την ε, εξωτερική πολιτική των χωρών μελών τη Ένωση. Επί του θέματο αυτού του Ισλαμικού κράτου και τη τρομοκρατία, δεν συμβαίνει αυτό ακριβώ με του Τούρκου φίλου. Τι γίνεται με τι διαβουλεύσει με την Τουρκία για το θέμα αυτό. Όχι για τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Και τρίτον, mm. εδώ μεταξύ μα, ω Ένωση, τι κάνουμε για να εναρμονίσουμε την ομοθεσία μας κατά της τρομοκρατίας. Η Γαλλία, όπως ξέρετε, προσπαθεί κάπως να συμμαζέψει την αντιτρομοκρατική της νομοθεσία για να βοηθήσει τη δικαστική εξουσία να ε, προσπαθεί να σταματήσει αυτούς που θέλουν να πάνε να γίνουν τζιχαντιστές. Αυτό όμως έχει έννοια μόνο αν όλες οι χώρες της Ένωσης έχουν ε, παρόμοια στρατηγική, παρόμοια νομοθεσία. Τώρα σε τι επίπεδο βέβαια θα γίνει ο συντονισμό είναι διακυβερνητικό θέμα, αλλά η υπηρεσία εξωτερική δράση και οι Κομισιόν προσπαθούν να ευνοήσουν αυτήν την σύγκληση και εναρμόνιση. Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τη Λιβύη όπου δυστυχώς ε, γίνεται αποτυχημένο κράτος όλο και περισσότερο και βεβαίω στι εκλογέ δεν υποστηρίχθηκαν πολύ οι Ισλαμιστικέ ομάδε, αλλά η βία του, οι θηριωδίε, οι εκτελέσει την προηγούμενη εβδομάδα ενό 19χρονου ε, blogger, όλα αυτά που γίνονται στην Τρίπολη, όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Λόγω του ότι αναπτύσσεται και το Ισλαμικό κράτο στην ε, Συρία και το Ιράκ. Μπορεί στη νότια γειτονία μας η Λιβύη να γίνει Ισλαμιστικό κράτος. Τι ρόλο παίζει το Σουδάν και το Κατάρ, θέλω να ρωτήσω. Ιδίω το Κατάρ, το οποίο έχει τεράστιε επενδύσει σε πολλά κράτη-μέλη τη Ένωση. Μεγάλη ζημιά κάνει γιατί του. Ε, είναι σχεδόν σίγουρο ότι του εξοπλίζει. Πρέπει να του ε, μαζέψουμε. Ξέρω ότι τα κράτη του Κολπέ έκανε ό,τι μπορούν. Αλλά μήπω μπορεί να κάνει την περισσότερη Ένωση. Συρία, Ιράν, Ιράκ τώρα. Είναι υπαρξιακή η απειλή που θέτει το Ισλαμικό κράτο για αυτή την περιοχή και οι περισσότερες μάχες γύρω από το κομπάνι γίνονται από κουρδικές δυνάμεις. Υπάρχει πρόθεση της Ένωσης να ξαναδεί τι καθεστώς δίνει στο ΠΚΚ ή το Συριακό αντίστοιχο YPJ που συμμετέχουν στις μάχες για να σταματήσουν το Ισλαμικό κράτος. Ιδιαίτερα γύρω από το Κομπάνι και για το ρόλο της Τουρκίας. Μετά την απελευθέρωση των 49 ομήρων, διπλωματών και άλλων που ε, είχαν απαχθεί στο, στη Μοσούλη θα κάνει η Τουρκία ό,τι μπορεί για να ιτηθεί το Ισλαμικό κράτο. Γιατί πριν από μερικά χρόνια λεγόταν ότι οι στρατιωτικέ δυνάμει και μυστικέ υπηρεσίε τη Τουρκία στήριζαν το Ισλαμικό κράτο και κάνουν τα στραβά μάτια. Όταν, έκαναν τα στραβά μάτια όταν ε, ξεκουράζονταν σε δικέ του περιοχέ για να γυρίσουν μετά πίσω να πολεμήσουν τον Ασάντ. Επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αναφερθώ τώρα στη Λιβύη, Συρία και Ιράκ, αλλά να εστιαστούμε πέρα των άλλο στην Λιβύη, γιατί πραγματικά δεν έχω δει πολλές φορές στη ζωή μου μια τέτοια τόσο βερμπαλιστική ε, δήλωση. Γίνονται τόσο πολλά στη χώρα. Έχουμε εδώ ένα ευχολόγιο. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, με τόσο γίνονται εκεί επί τόπου. Μα τι είναι αυτό, κάποιο είδου ε, προσευχή. Ο ρόλος των γυναικών για, την, ε, για το μετασχηματισμό κλπ. Όλα αυτά είναι άσχετα με την πραγματικότητα. Και επίσης, άλλο παράδειγμα, στο σημείο 14 που λέει για την αύξηση του λαθρεμπορίου όπλων. Όποιο ξέρει δύο πράγματα για τη Λιβύη, ξέρει ότι εξάγει όπλα η Λιβύη, δεν εισάγει. Και Σούφραγκα, Τρούν, Μουρσούκου, Άουελ Κιμπίρ, στο, στο νότο δηλαδή τη χώρα ή στη Σέμπχα, εκεί έχουμε μια μπαρουταποθήκη τεράστια ε, σε σχέση και με, και με το Νταρφούρ, του Σουδάν δηλαδή. Και φεύγουν από εκεί όπλα για Νιγηρία, ε, Νταρφούρ, Μαλή και τελικά ποιος φταίει. Φταίνε αυτοί οι λαθρέμποροι όπλων. Οπότε ε, συμπαθάτε με, αλλά από αυτό το κείμενο προκύπτει ότι δεν έχετε την και το τι γίνεται εκεί. Δεν έχει κυβέρνηση η χώρα. Είναι εικονική η κυβέρνηση. Μια βιτρίνα. Στο, το Μπρουκ έχουν πάει και μερικοί εκεί. Τους προστατεύει ο Χαλίφης Χάφτερ. Και υπάρχει άλλη κυβέρνηση ε, στην ε, Τρίπολη με ένα κοινοβούλιο. Όμως ε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ε, με την πραγματικό για την πραγματικότητα εκεί ε, και από διπλωματικές περιοχές. Τελικά δηλαδή εκεί υπάρχουν κάποιοι, κάποιες ε, φυλές, ομάδες, ο, ο καθένας φροντίζει τα συμφέροντά του και όλοι μαζί διέπονται από τους οπλαρχηγούς και αυτό εδώ το, το, κείμενο δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα δύο τρίτα του νότου της χώρας εκεί είναι, όλα, είναι, είναι για όλα τα συμφέροντα, για τα λαθρεμπόρια ε, και το, το Τσάδ, η Νιγηρία, ε, οι έμποροι τα συμφέροντα από εκεί περνάνε. Είναι ένας ε, κεντρικός διάδρομος που αφορά τη ζώνη του Μπορκού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά γιατί αυτό πάει να πει ότι στην, στην Νιγηρία, η Μπόκο Χαράμ συνδέεται με την τρομοκρατία σε άλλα μέρη της περιοχής. Θυμάστε τότε που είχαν ε, απάγει ε, εκατοντάδες ε, κοριτσιών ανηλίκων. Πού είναι όλα αυτά εδώ στο κείμενο. Εδώ λέμε ότι θα πρέπει τα οι εμπλεκόμενοι να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. για να κάτσουν θα πρέπει να του ενδιαφέρει, να έχουν συμφέρον να κάτσουν, να συνοηθούν. Μα εκεί έχουμε συμφέρον τα λεφτά και τι εξαγωγέ πετρελαίου. Αυτά όλα είναι εκπληκτικά. Να περιμένουμε η κυβέρνηση τη Λιβύη να σταματήσει της ε, εξαγωγή του πετρελαίου. Ε, είναι σαν να εύχεται κανείς, σαν να θέλει κανείς να ξεράνει τον ωκεανό. Μα έχουμε αυτές τις εμπορικές ροές, αυτές τις εξαγωγές. Και όσον αφορά το Ισλαμικό κράτος, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι έλεγχος και κυρώσει για ε, όλες αυτές τις χιλιάδες κινήσεων μεταφορών που γίνονται από την Τουρκία. Περνάνε από εκεί μέσα οι λαθρέμποροι και γίνεται λαθρεμπόριο στο Κουρδιστάν. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι απλό, γιατί πρόκειται για χιλιάδες ε, φορτηγών. Όσον αφορά τι εξαγγελίες πετρελαίου, ε, υπάρχουν εκεί κάποιοι παραστρατιωτικοί που το ελέγχουν και με τους ε, σωλήνους με τους αγωγούς που μεταφέρουν το πετρέλαιο. Ναι, ναι, κλείνω, κλείνω πρόεδρε. Πρόεδρος. Κύριε, συνάδελφε. Τώρα, το πρωί μιλήσατε 10 λεπτά και τώρα άλλα 5. πώ πώς θα μιλήσουν οι άλλοι. Ναι, ναι, ναι, κλείνω. Άρα θα πρέπει άπαξ και ε, διαπαντός να κλείσουμε τον αγωγό πετρελαίου, την κάνουλα. Κυρία Αλιώτα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά αυτά τα δύο θεματάκια. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την Λιβύη, έχουν τους ανταγωνισμούς μεταξύ της Κυριναϊκής, ε, της Τρίπολης και των φυλών του Νότου, το οποίο ανάγεται στο μακρινό παρελθόν, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η βάση του, του, προβλήματος είναι η, η άνηση κατανομή του πλούτου και συγκεκριμένα του πλούτου από το πετρέλαιο διότι πέραν όλων που θα μπορούσε να πει κανείς για όλες τις άλλες αντιπαραθέσεις, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Τώρα, τι προτείνουμε, εάν θέλουμε πραγματικά να παρεύουμε ούτως ώστε να ρυθμίσουμε την κατάσταση. Επίσης, για Ιράκ και Συρία, συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτού του είδους ε, ε, η απομόνωση, να μην υπάρχει πρόσβαση στα όπλα, και να μην έρχονται από τις χώρες μας εκεί πηγαίνουν τζιχαντιστές. Όμως ε, θα πρέπει και να τους απομονώσουμε από την αραβική κοινή γνώμη. Να μην ξεχνάτε ότι οι συγκρούσεις εκεί ε, ε, είναι κάτι το οποίο το πήρε πάρα πολύ και η Χαμάς, αλλά και το ότι ολένα και περισσότερο οι ηγέτες των εκεί χωρών ε, προέρχονται από το λαό, τελο πάντων λαμβανουν υπόψη τη γνώμη του λαού. Άρα είναι απαραίτητο αυτό ότι να είμαστε πιο ανοιχτοί από ό,τι σήμερα και όλα τα κράτη, όχι μόνο η Τουρκία αλλά και οι πιο μακρινές αραβικές χώρες, να συμμετάσχουν, να καταδικάσουν, να αναλάβουν δράση. Και μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό για μας και για το μέλλον να αντιπαραθέσουμε τους Μητροπαθείς Μουσουλμάνους στους ε, Ισλαμίστες, στους ακραίους. Τα πράγματα θα έχουν μια μακρά πορεία και άρα εμείς θα πρέπει στην παρέμβασή μας να προσέξουμε, να κάνουμε προσεκτική διάκριση μεταξύ εξτρεμιστών, ε, τρομοκρατών και από την των μετριοπαθών. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Σας προτείνω να, οι υπόλοιποι να λάβετε το χώρο όταν ε, συζητήσουμε την υπόλοιπη Δεν το απόγευμα. Συζητείτε γιατί ήδη μας έχουμε αργήσει. Λόζιν, Καστάλτο και οι άλλοι. Να είστε οι πρώτοι που θα λάβετε το λόγο στη συνεδρίαση που κάνουμε στις 3. Και σας ευχαριστώ. Ε, μερικοί από σας, ελάτε. Μην με αφήσετε μόνο με τον κύριο Γκρέσλε. Yeah. Τι φοβάστε, ε, βέβαια.